Ευρωπαϊκή Αριστεράς μου ζητά να ονομάσω την κυρία ε, Στεφανία Τόρε Μαρτίνο στη θέση του κυρίου Παύλου Ετσενίκε ω μέλους τη επιτροπή περιβάλλοντο Δημόσιας Υγείας και ασφάλεια των Τροφίμων και μέλο αντιπροσωπείας για τι σχέσει με την Λαϊκή Δημοκρατία τη Κίνα. Υπάρχουν αντιρρήσει. Εγκρίνεται.